Χθε, αγαπητοί συνάδελφοι, μια τρομοκρατική επίθεση έπληξε χθε την Τινησία, την πρωτεύουσα της Τινησίας. 14 μέλη της Προεδρικής Φρουράς χάσαν τη ζωή τους. Εξ ονόματος λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου